συζήτηση με τη δήλωση της Επιτροπής. Κύριε Ντεγκούχτ, έχετε το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, uh, Madam President. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, η Ευρώπη προβληματίζεται βαθιά από τις συνέβη καταστροφικές των πλημμυρών στο Πακιστάν που κατέψαν τις ζωές και τις περιουσίες πάντως σε όλη τη χώρα. Η καταστροφή αυτή έχει κλίμακα χωρίς προηγούμενο και πάρα πολλές δαπάνες χρειάζονται ε, γιατί ήδη η οικονομία ήταν ευάλωτη, χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, ήταν πάρα πολύ σοβαρή αυτή η κρίση, άρα χρειάζεται άμεση απόκριση και επίσης θα πρέπει να πάρουμε υπόψη την στρατηγική σημασία της ε, χώρας αυτής όσον αφορά την ανάπτυξη, όσον αφορά την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στις 16 Ενάτου το Συμβούλιο ε, ε, απίθυνη έκκληση ώστε να έχουμε κάποια μέτρα μακράς και βραχίας ε, πνοής ούτως ώστε να βοηθήσουν το Πακιστάν και ήταν γενναιόδορη και άμεση η απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι έχουμε εισφέρει ε, στην προσπάθεια αυτήν κατά 320 εκατομμύρια ευρώ τα κρατημέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε είδος και σε χρήματα βοήθησε δηλαδή πάνω από το 60% της όλης βοήθειας ε, από πλευράς της παγκόσμιας κοινότητας ε, αναγνώρισε το Συμβούλιο ότι εκτός από όλα αυτά χρειάζεται βοήθεια, χρειάζονται εμπορικά μέτρα για να βοηθήσουμε την ανασυγκρότηση την οικονομική της χώρας. Γιατί το εμπόριο είναι μέρος αυτής της ε, απόκρισης που πρέπει να δώσουμε στην κρίση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 7 Δεκάτου μονομερός να παγώσει τους εισαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα από το Αφγανιστάν. Και ε, αυτή μας την πρόταση σας υποβάλλουμε. Οι 75 ε, τέτοιους δασμούς θέλουμε να παγώσουμε που αντιστοιχούν στο 27% των εμπορικών ροών του Πακιστάν προς την ΕΕ του που αντιστοιχεί σε ένα ποσό 900 εκατομμυρίων. Ε, αυτό αντιστοιχεί σε 100 εκατομμύρια ευρώ εισαγωγών του Πακιστάν. Έτσι θα βοηθήσουμε μέσω πρόθεσμα στην ανασυγκρότηση της χώρας. Σε συνέπεια όλων αυτών θα βοηθήσουμε ε, ε τη, χώρα αυτή, θα κρατήσουμε αυτά τα μέτρα δύο χρόνια και θα πρέπει να δούμε ότι τα φαντουργικά είναι 60% των εξαγωγών και έχουν προταθεί μέτρα απορρίθμισης για αυτά τα προϊόντα της κλωστοφαντουργίας. Έχουμε και άλλα προϊόντα, εθανόλη, Φερρυπίν και αυτά θα καλυφθούν από αυτές τις απαλλαγές ή στους δασμούς. Ελπίζουμε επομένως να, τα, τα μέτρα αυτά να αρχίσουν να ισχύουν από 1η Πρώτου 2011. Και επίσης συνεργαζόμαστε με διάφορα άλλα μέλη του ΠΟΕ, γιατί θα πρέπει να υπάρχει το πράσινο φως από τον ΠΟΕ πριν ε, τρέξουν αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει όλα αυτά επομένως να υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη και τις ευαισθησίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιομηχανικά θέματα και για αυτό και προτείναμε και εμεί αντιστοίχω να ληφθούν υπόψη αυτέ τι ευαισθησίες, ιδίω όσον αφορά την κλωστοεφαντουργία. Έγινε κάποια ανάλυση και είδαμε ότι οι συνέπειε δεν θα είναι τρομερές στην παραγωγή μας. Είπαμε για τις εισαγωγές των 100 εκατομμυρίων του Πακιστάν από την Ένωση και είναι 0,5% ε, της παραγωγής της δικής μας όσον αφορά τα απορριθμισμένα ούτως ε, αυτά τα προϊόντα γιατί το σύνολο της παραγωγής είναι 24 δισεκατομμύρια και επομένως ελπίζουμε ότι θα ευδοκιμήσει αυτή η πρόταση γιατί έτσι θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το ψηφιδωτό Τη ανθρωπιστική μας βοήθειας, μια που οι ανάγκε της χώρας αυτής είναι χωρί προηγούμενο στην ιστορία. Το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό. Και μπορείτε να υπολογίζετε στι ε, προσπάθειες της δικές μου αλλά και του, του των συνεργατών μου ε, σε ό,τι ε, χρειάζεστε. Τώρα το λόγο θα πάρουν ομιλητέ εξ των πολιτικών ομάδων για το... παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μιλούμε για την κατάσταση στο Πακιστάν. Οφείλω να σας πω ότι η κατάσταση της χώρας αυτής είναι τραγική για την Ευρώπη, αλλά επίσης και για όλες τις χώρες που έχουν δυσκολίε όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Να ένα παράδειγμα, η κλωστοϊφαντουργία είναι το 11% των εξαγωγών της χώρας μου της Πορτογαλίας. 22% της απασχόλησης η μεταποίηση και βιομηχανία. Και επίσης η κλωστοφαντουργία ε, είναι 80% ε, διαφόρων άλλων κλάδων. Δηλαδή Ίσως για άλλες χώρες της Ένωσης αυτό δεν πάει να πει πολλά πράγματα, αλλά για μας είναι τερατώδες. Γι' αυτό και θα πρέπει να απαιτηθούν ε, μέτρα σκληρά, μέτρα ούτως ώστε να ε, τυθασευτούν τα δημοσιονομικά αλλά και ε, το δημόσιο χρέος. Όμως Παράλληλα με τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται, δεν είναι δυνατόν να θέτουμε ένα αμφιβόλο την παραγωγή, να θέτουμε ένα αμφιβόλο θέσει απασχόληση στι χώρε μα. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία αποτελεί μια αντίφαση στην ε, λογική της αγοράς. Ε, δεν είμαι υπέρ του προστατευτισμού, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, μια αγορά η οποία λειτουργεί με δίκαιους όρους και είναι υγιής. Έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα του Πακιστάν, τα οποία παράγονται πολύ πιο φτηνά από ό,τι τα αντίστοιχα δικά μας, γιατί φυσικά οι προδιαγραφές εκεί είναι με, με τον πύχη πολύ πιο ε, χαμηλά. Όλα αυτά τι είναι, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει γενικό κόστος, δεν υπάρχει κανένα είδους πρόνοια για τους εργαζόμενους στο Πακιστάν, κανένα είδους κοινωνική προστασία και για το περιβάλλον. Καμία σχέση δεν έχουν με τα δικά μας προβλήματα για την εργασία των ανηλίκων. Δεν του νοιάζει. Ούτε έχουν τίποτε νομοθεσία, νόμους και νομοθεσίες για, για τις πρώτες ύλες και για την υγιεινή στο χώρο εργασίας. Άρα θα πρέπει να καταλάβετε το ότι αυτή τη στιγμή ε, χρειάζεται μια σοβαρή έκθεση που να ζυγίζει τις συνέπειες για τα κράτη-μέλη. Ήδη μπορούμε να προβλέψουμε τις συνέπειες ή κάποιες από αυτές. Πάμε για πτώχευση βιομηχανιών και επιχειρήσεων στην Πορτογαλία. Πάμε για ανεργία και αυτό θα πρέπει να το πούμε και κάποιος θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες για όλα αυτά. Ξέρω ότι αυτή η πρόταση θα πάρει το δρόμο της, αλλά τουλάχιστον ας ε, προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ε, συνέπειες ή τουλάχιστον να κάνουμε κάτι για την εθανόλη. Προβλέπονται κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί. Επίσης όσον αφορά τις προσωρινές ενισχύσεις να το εξετάσουμε και αυτό. Είναι αδύνατη η, η αναμέτρησή μας, ο ανταγωνισμός μας με τις επιχειρήσεις της ε, πακιστανικές χωρίς καμία ενίσχυση. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μάρτιν εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Εγώ έχω κατανόηση για τα όσα λέει ο κύριος Μέλλο, αλλά δεν συμφωνώ. Εγώ χαίρομαι για την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταργηθούν οι του Πακιστάν. αυτή η χώρα περνά από δυσχερέστατη ε, περίοδο Γνωρίζουμε για τι πλημμύρε, γνωρίζουμε για το κόστο ε, του αγώνα κατά των Ταλιμπάν που, έχει, φτάσει στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα και ε, ούτω καθεξή. Ε, όλα αυτά αποτελούν βαρύτατα πλήγματα για οποιαδήποτε χώρα. Αυτό που με ικανοποιεί στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι προσφέρουμε τη δυνατότητα στο Πακιστάν να αντεπεξέλθει στι δυσκολίε του μέσω του εμπορίου είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 75, ε, είδη προϊόντων που δεν θα αποτελέσουν ε, σημαντική ζημιά για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή βιομηχανία και ίσως μάλιστα δεν, ε, ακόμα καλύτερα μάλιστα, δεν θα βλάψουν τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ανταγωνισμό με το Πακιστάν. Αυτά είναι θετικά. Το δεύτερο που βρίσκω λογικό ε, στοιχείο στην πρόταση της Επιτροπής είναι ότι έχει περιορισμό χρόνου και δεν γίνεται μια μονομερής ε, προσπάθεια και ζητείται από το Πακιστάν να ευθυγραμμιστεί με τις κοινωνικές ε, προδιαγραφές μέχρι το 2014 ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στο GSP Plus μέχρι το 2014. Ταυτόχρονα λοιπόν δεν δίνει λευκή επιταγή στην, ε, επιταγή στην ε, ε, πακιστανική κυβέρνηση. Τους λέει εάν θέλετε να συνεχίσετε να αποφελείστε από, ε, αυτές, από αυτά τα πλεονεκτήματα θα πρέπει να καταβάλλετε μια προσπάθεια. Βρίσκω ότι αυτή είναι μια σωστή και γενναιόδορη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάρει ο κύριος εκ μέρους Συμμαχίας των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επιτροπή. Η σημερινή συζήτηση είναι ένα σημείο που συναντώνται δύο βασικέ αρχέ. Από τη μία πλευρά η υποχρέωση τη αλληλεγγύη σε μια χώρα που πλήγει από μια φυσική καταστροφή. Από την άλλη η ανάγκη για μια εμπορική πολιτική που να είναι εξισορροπημένη. Με την πρόταση της ετροπής για μια άρση των δασμών στο Πακιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά αποφεύγει μια πολιτική απλής παροχής βοήθειας, επιτρέποντας στο Πακιστάν να ενισχύσει την οικονομία και την κοινωνία του. Και η 78 ε, τέσσερις κατηγορίες ανήκουν στον τομέα της ένδυσης και της κλωτοφεντουργίας. Αυτό είναι απόφευκτο για μια χώρα που αυτό που εξάγει στην ουσία έχει να κάνει με την ένδυση και την κλωστοφαντουργία. Ε, οι, εμείς οι ελεύθεροι δημοκράτες προτιμάμε αυτό από την ανθρωπιστική βοήθεια γιατί αυτό θα οδηγήσει τη χώρα σε μια ανάκαψη. Παρόλα αυτά θα πρέπει, όπως θύμισε ο συνάδελφος μέλο προηγουμένως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς. Ο Επίτροπος γνωρίζει καλά την κρίσιμη κατάσταση σε ορισμένους τομείς της κλωστοφαντουργίας η περίπτωση του Πράτο. Το Πράτο είναι ένα θέμα που θίξαμε και σήμερα το απόγευμα. Ξέρετε ότι είναι μια κατάσταση που ετέθη εκτό ελέγχου από τι εθνικέ αρχέ. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί, αναπτύσσονται πάρα πολλέ παράνομε δραστηριότητε. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε μόνον από την Ευρωπαϊκή Κλωστοφαντουργία να πληρώσει το τίμημα τη ε, αλληλεγγύη μα στο Πακιστάν. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε τρία πράγματα. Καταρχά, κανονισμού για να αποφευθεί τη δημιουργία τριγώνων με άλλες χώρες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τους θετικούς φόρους του Πάκισταν, να μην επιδεινώσουμε την κρίση της ευρωπαϊκής ε, κλωστοφαντουργίας ε, μέσα από μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια στήριξη, για παράδειγμα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο για άλλες χώρες ε, που ενδεχομένως θα πληγούν από παρεμφερείς φυσικές καταστροφές. Με αυτόν τον τρόπο η βοήθεια προς το Πακιστάν πιστεύω ότι θα μας βρει όλους σύμφωνους ακόμα και μακροπρόθεσμα. Και βεβαίως η βιώσιμη βοήθεια είναι αυτό που χρειάζεται αυτή η χώρα. Προσέχετε να μην ξεφεύγετε κύριοι συνάδελφοι. Τώρα ε, για τους Ευρωπαίους συντηρητικού, ο κύριος Βλοζόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Επίτροπε. Σήμερα οφείλουμε να συζητήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βοηθήσουμε το Πακιστάν να ξεπεράσει τις συνέπειες αυτής της πλημμύρας. 14 εκατομμύρια υποφέρουν από αυτή την βιβλική καταστροφή. και οι ηλικίες καταστροφές εκεί είναι τεράστιες και θα υπάρξουν ε, συνέπειες λόγω του ότι το Πακιστάν είναι πάρα πολύ βασικός παραγωγός βαμβακιού. Η παραγωγή επομένω θα συρρυκνωθεί όπω συρρυκνώθηκε και η σοδιά και ήδη οι παραγωγοί επεφάσισαν ότι θα ανέβει η τιμή, η τιμή του βαμβακιού, η τιμή των κλωστοφαντουργικών γενικότερα. Ξέρετε, εκτός από τα ρούχα, το μπαμπάκι χρησιμοποιείται και για πάρα πολλά άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Επομένως, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο. Μέρο τη ενωτική αριστερά. Numa mão, nós temos grandes importadores europeus. Και, κυρία Πρόεδρε, από τη μία μεριά έχουμε κάποιου Ευρωπαίου εισαγωγεί που κερδίζουν ένα σωρό λεφτά από τι εισαγωγέ που από το Πακιστάν. Από την άλλη μεριά όμω έχουμε πάλι κάποιου ε, κλωστοεφαντουργού Πακιστανού οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε κάποιε περιοχέ που δεν χτυπήθηκαν την καταστροφή. Επομένω, με αυτή την πρόταση τη Κομισιόν αυτοί πρόκειται να ε, πλουτίσουν αδικαιολόγητα. Διότι με αυτή την πρότασή σας ε, κύριε Επίτροπε ούτε οι γέροι ούτε τα παιδιά ούτε οι άστεγοι δεν θα ωφεληθούν. Θα κερδίσουν οι πλούσιοι επιχειρηματίες. Αυτό το οποίο κάνετε τώρα είναι το να χρησιμοποιείτε σαν μέσο την καταστροφή και ε, τις θεομηνίες για να μπορέσετε να κλείσετε κάποιες ε, παχυλές συμφωνίες. Γι' αυτό και θεωρώ απαράδεκτη την πρόταση της Κομισιόν. κύριε Πόρτας. Τώρα για την Ευρώπη τη ελευθερία και τη Δημοκρατία, για 1,5 λεπτό, ο κύριος Ντάρκμουντ θα πάρει το λόγο. Στο παρελθόν έχω επικρίνει κατ' επανάληψη τον Πρωθυπουργό τη μεγάλη Βρετανία, κύριο Κάμερον. Ωστόσο, ήταν σωστό αυτό που έκανε, ότι ζήτησε δηλαδή εμπορικές προτιμήσεις υπέρ του Πακιστάν. Εγώ λέγω ζήτησε, διότι ακριβώς αυτό έπρεπε να πράξει. Από τις ένταξεις του στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της, ε, του κόσμου, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει η δική του κυρίαρχη εμπορική πολιτική, ούτε καν μέσα στα πλαίσια της κοινοπολιτείας. Ωστόσο είναι προ το συμφέρον και του Ηνωμένου Βασιλείου να αποκτήσει εμπορικέ προτιμήσει το Πακιστάν. Σπάνια συμφωνώ με τον Ντέβιτ Μάρτιν, αλλά συμφωνώ επί του προκειμένου. Το Πακιστάν είναι και αναπτυσσόμενη χώρα με 170 εκατομμύρια πληθυσμό και με στατηγικά σύνορα με το Αφγανιστάν, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια χώρα η οποία διαθέτει 30 πυρηνικέ κεφαλές. Οι επιπλοκές στην ασφάλεια μιας ενδεχόμενης κατάρρευσης του πακιστανικού κράτους θα ήταν καταστροφικές για την ασφάλεια ολόκληρου του αναπτυσσόμενου, του αναπτυγμένου μάλλον ε, κόσμου. Οι εμπορικές προτιμήσεις λοιπόν υπέρ του Πακιστάν ίσως να συμβάλλουν στην αναχέτηση ενός τέτοιου ενδεχομένου. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Κάσπαρη για τρία λεπτά. Three minutes. Yeah, Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας θυμηθούμε όλοι πόσο δραματική ήταν η κατάσταση του Πακιστάν προ λίγων εβδομάδων. Ολόκληρα τμήματα της χώρας βρίσκονται ακόμα κάτω από τα νερά. Περιοχές της χώρας που είναι μεγαλύτεροι από πολλές δικές μας χώρες μέλη. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν βαρύτατα προβλήματα, νοσοκομεία, παιδική σταθμή έχουν καταστραφεί, σχολεία και ούτω είναι πραγματικά μια κατάσταση αδιανόητη. Ωστόσο όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Το πρόβλημα, όπως λέμε εμείς, είναι πώς να το κάνουμε χωρίς να προκαλέσουμε ζημίες αλλού. Η άμεση ε, οικονομική ενίσχυση θα είχε επιπτώσει στον προπολογισμό μας. Η ε, ενίσχυση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εμπορικές προτιμήσεις και εδώ ορισμένοι εκφράζουν επιφυλάξεις γιατί ενδέχεται να πληγούν οι δικές τους βιομηχανίες η ε, Κομισιόν δεν προτείνει χρήση του γενικού συστήματος προτιμήσεων. Εγώ το βρίσκω σωστό. Και η πορεία μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου βρίσκω ότι είναι σωστή. Δηλαδή βοηθούμε το Πακιστάν να βοηθήσει τον εαυτό του στην ουσία. Όμω μένουν ακόμα πολλά ερωτήματα ανοιχτά σε ό,τι αφορά τι ενδεχόμενε επιπτώσει για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εξετάζοντα το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόταση δηλαδή κανονισμού, στην αρχή διαλαμβάνεται ότι οι τιμέ ότι οι επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη μεριά θα είναι απώλεια 80 εκατομμύρια ευρώ για τον δικό μας προϋπολογισμό. Θα χάσουμε δηλαδή συνολικά δασμούς ε, της τάξης των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ θα προτιμούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προσφέρει πλήρης πληροφορίες. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι πρέπει να βοηθήσουμε το Πακιστάν. Και είμαι διατεθειμένο να βγω και να εξηγήσω στου Ευρωπαίου πολίτε και στου ψηφοφόρου μου τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή. Είμαι όμω πεπισμένος, κύριε Επίτροπε, ότι σήμερα θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σα δίνεται ενώπιον μα, αλλά και στι επόμενε εβδομάδε. αφενό να πείστε του ευρωβουλευτέ ότι τα μέτρα σα είναι σκόπιμα και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία που σας δίνετε να καταδείξετε και άλλους δρόμους για να ενισχύσετε βιομηχανίες όπως της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών να ε, σταθούν καλύτερα στα πόδια, στα τους. Έτσι νομίζω σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες θα επιτύχετε πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της προτάσεώς Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάσπαρη. Ο κύριος Σούστα τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση της κρίσης που διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη. Κρίση που αφορά την ανάπτυξη, την εργασία, την απασχόληση. Ειλικρινά αναρωτιέμαι ποια είναι η λογική που συχνά εμπνέει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ιδιαίτερα την Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις. Αυτή η διάταξη και είναι μια διάταξη της Επιτροπής, ένα μέτρο της Επιτροπής που θα θυσιάσει πολλούς βιομηχανικούς τομείς, ιδιαίτερα τον τομέα της κλωστοφαντουργίας. Και αναρωτιόμαστε γιατί σε ένα πλαίσιο όπως το παρόν θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα κάποιος ε, λέει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο του να θέλει να παίξει η Ευρώπη πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις. Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία σχέση ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ευρώπης. Πολύ μικρότερο ρόλο παίζει προσπάθεια να μειωθεί μεταξύ των άλλων και η τρομοκρατική πίεση στο εσωτερικό ορισμένων συστημάτων ή που ενεργοποιείται από ορισμένα πολιτικά και θεσμικά συστήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση σχέση, δεν έχουν καμία σχέση ούτε οι πρόσφατες πλημμύρες ε, γιατί δεν έχουν πληγεί οι κλωστοφαντουργικές περιοχές. Ο βασικός λόγος είναι ότι θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε έναν τομέα ε, και αυτό υπέρ των μεγάλων ε, δικτύων διαδομής για να πλήξουμε την μεταβλητική βιομηχανία που βρίσκεται σε ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε. Και αυτό είναι λάθο από την άποψη τη ανάπτυξη, τη εργασία, τη απασχόληση σε μια στιγμή σοβαρή οικονομική κρίση και στιγμή ανάγκη για πραγματική ανάπτυξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση των εξαγωγών στα, μέσα στι μεγάλε αγορέ. για λεπτά λόγο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τους συναδέλφους Μάρτιν και Τεσκάσπερη για τα τόσο χρήσιμα σχόλιά τους. Μετά από τις πλημμύρες στο Πακιστάν, κυρία Πρόεδρε, επισκέφθηκα τη χώρα για να δω μόνο μου, μόνος μου την έκταση της καταστροφής. Η καταστροφή που έχει προκληθεί από τις πλημμύρες είναι η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία του Πακιστάν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινο. Όταν συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν στις 27 Σεπτεμβρίου, έδειξε να εκτιμά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χαρακτήρισε θαραλέα. Ήταν θαραλέος ο τρόπος που όπως περιγράφει από τον Επίτροπο. Θα πρέπει να έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι συνεχίζουμε να αντιδρούμε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Η Επιτροπή συμφώνησε με την νομοθετική πρόταση να μειωθούν σε μηδέν οι φόροι επί 74 ε, προϊόντων. Και αυτό θα προωθήσει τι εξαγωγέ του Πακιστάν κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι μία ε, δοκιμή της αξιοπιστίας ε, της ε, Επιτροπής. Θα πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι μεταφράζεται η πολιτική συμφωνία σε δράση, έτσι ώστε να γίνει μια πραγματική διαφορά και να αποκτήσει ή να δώσουμε μια νέα πνοή ζωής στο Πακιστάν. Σε τελευταία ανάλυση είμαστε ο μεγαλύτερο εταίρο τους. Καταλαβαίνω ότι τους προβληματισμούς του συναδέλφων. Είναι σωστό αυτό να δώσουμε σωστές απαντήσεις, να είμαστε δίκαιοι αλλά φιλόδοξοι. Οι εκχωρήσεις θα πρέπει να δείξουν μια αξιόπιστη προσπάθεια από πλευρά της Ευρώπης και να συνεπάγονται συγκεκριμένα ωφέλη ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξουμε ότι συνυπολογίζουμε την επίπτωση που θα έχει και σε εμά και στι λιγότερο ευδημένες χώρε. Μέσα από αυτή την πρόταση πιστεύω ότι φαινόμαστε φιλόδοξοι, φαινόμαστε θαραλέοι αλλά κυρίω είμαστε δίκαιοι απέναντι στον εαυτό μα, αλλά και απέναντι στο λαό του Πακιστάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρύμ. Ο κύριος Χίγινγκς έχει το για ένα Κύριε Πρόεδρε, έχουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν πληγεί και αυτοί χρειάζονται άμεσα βοήθεια. Κάτω είναι οι ανήλικοι που είναι άστεγοι, είναι να πεθάνουν από πείνα. Και πάρα πολλά εκατομμύρια γεωργών και εκεί εκτιμώνουν τώρα ε, είναι, στο έλεος των ε, γεωκτημόνων. Χρειάζεται επομένω να του βοηθήσουμε με λοιπάσματα και όλα τα άλλα, ούτω ώστε να μπορέσουν να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά του και να υπάρχει παραγωγή τροφίμων. Όμω θα πρέπει να γίνει αναδιανομή τη γη. Θα πρέπει αυτοί οι, ε, οι ακτήμονε να αποκτήσουν κάποια κτήματα. Και αυτά τα, τα, τα ξέρουμε στην ε, Ιρλανδία πως έγιναν και χρειάζεται επομένως να βοηθήσουμε όχι τους γεωκτήμονες αλλά τους ε, φτωχούς, ούτε τους βιομήχανες, αλλά αυτούς που θα ωφεληθούν αν υπάρχουν δίκαιες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα. Προσοχή να μην βοηθήσουμε στις αγορές των εμπορευμάτων τους ε, κερδοσκόπους. Ε, Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, όλους μας απασχολούν οι ε, πλημμύρες στο Πακιστάν και οι επιπτώσεις που έχουν στην οικονομία του. Μας απασχολούν όμως παράλληλα και η πρόταση της Επιτροπής μολονότι ε, το ερέθισμα το έδωσαν οι πιαυλίες κρατών και κυβερνήσεων. Ο κανονισμός προτείνεται από την Επιτροπή επικεντρώνεται συνήθως στην εξαίρεση από τους δασμούς στον τομέα της βριστοδεψίας και της κλωστοφαντουργίας που είναι το 60% των εξαγωγών του Πακιστάν με ένα τζίρο περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον κλωστοφαντουργικό τομέα και 510 εκατομμύρια ευρώ <coughs> για τη βριστοδεψία. και αυτό σε περιοχές που δεν έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Οι πολιτικές ενδείξεις αφορούν στην επιλογή μια στοχοχευμένη βοήθεια που δεν ε, θα πλήξει το μη της ευρωπαϊκή οικονομία. Η άρση των φόρων θα έχει άμεσε επιπτώσει στην κλωστοφαργική βιομηχανία και στη βιοξοδεψία τη Ευρώπη και, και θα χαθούν πάρα πολλέ θέσει εργασία τα τρία χρόνια που προβλέπεται από τον κανονισμό. Αυτά τα μέτρα θα επιβαρυνθούν από το σύστημα γενικευμένων ε, δασμολογικών προτιμήσεων που θα επεκταθεί το 2013 και στο Πακιστάν. Κύριε Κύριε, ε, κύριε Επίτροπε, έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι υιοθετούνται οι ε, έκτακτα μέτρα γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε μια φτωχή μεγάλη χώρα επειδή επλήγει από μια κρίση η οποία επιδεινώνεται και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και στο ότι δεν έχει προσαρμοστεί στους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργάνωση Εμπορίου που ευνοούν χώρε όπω η Κίνα και η Ινδία σε σχέση με πιο φτωχέ χώρε. Τα κατεξαίρεση μέτρα που βοηθάν μια χώρα δεν μπορούν να συνεπάγονται κρίση για άλλε χώρε. Η πρόταση τη Επιτροπή κατά συνέβεια θα πρέπει να είναι διορθωτική και κατά συνέπεια θα πρέπει να την απασχολήσει και η να την εξαχωσχολήσουν και οι εξαγωγέ του Πακιστάν και να ληφθούν τη σοβαρά υπόψη το θέμα του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και τη καταπολέμηση τη τροποκρατία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε το Πακιστάν, αλλά μέσα από σαφεί συμφωνίε στα πλαίσια του πλήρου σεβασμού τη πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Η κυρία Ανδρέα Μπαρέα έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι πλημμύρες Ιουλίου και Αυγούστου φέτος ε, είχαν σαν αποτέλεσμα 20 εκατομμύρια πλήγησαν 1.800 νεκρούς και πάρα πολλοί, περισσότερο αυτούς χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και επομένω θα πρέπει όπως μας είπατε αυτά τα 20 εκατομμύρια να τα δώσουμε, εμείς ε, δώσαμε 11 εκατομμύρια ως ε, Ισπανία. Δεν μιλάμε για εμπορική συμφωνία, μιλάμε για στρατηγική ανάπτυξη της ε, χώρας. Και εσείς με την εντολή του Συμβουλίου αυτά τα 75 προϊόντα για μια τριετία τα απελευθρώσετε από δασμού, όπω είπε το Συμβούλιο, και επομένω θα πρέπει να δούμε πώ οι εξαγωγέ του, του, Πακιστάν θα, θα έχουν κάποιε συνέπειε στην Ευρώπη ε, Τέτοιε συνέπειε που θα τι θυσιάσουν λαμβάνοντα υπόψη την ιδιορυθμία κάθε χώρα η εθανόλη, τα κλωτεφαντουργικά και τα δερμάτινα είδη, να δούμε τι θα γίνει με αυτούς του καταλόγους των προϊόντων ε, που πρέπει να τι προσέξετε γιατί θα έρχονται σε σύγκρουση με ε, αυτά που είπατε. 16% είναι η δική μας η συμβολή σε αυτά, 16% είναι τα κλωστοφαντουργικά στην Βαλένθια ε, από το σύνολο της χώρας και γιατί η αγορά αυτή στην Βαλένθια ε, είναι πάρα πολύ σημαντική όπως και η Γερμανία όπως και η Γαλλία και αυτό μας χτυπάει την αγορά οι εισαγωγές δηλαδή από το Πακιστάν γι' αυτό και θα πρέπει να σας πω ότι οφείλετε να κάνετε μια στρατηγική μελέτη και θα πρέπει να ε, ζυγίσετε τις δυνατότητες του Πακιστάν να γίνει μια ετήσια αξιολόγηση των συνεπειών της συμφωνίας που μας προτείνεται. Ο κύριος Φέρνερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η βοήθεια προς το Πακιστάν μετά τις καταστροφές που προήρθαν από τις πλημμύρες μας ευρίσκει σύμφωνους Χαίρομαι που αντιδρά με ταχύτητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντας μέτρα. Βέβαια, αυτά ε, συνεπάγονται κάποιες δαπάνες. Αλλά τι ρόλο παίζουν αυτές. Θα κοστίσει χρήματα. Βέβαια, με την έκπτωση των δασμών η βοήθεια αυτή. Βεβαίως, πρέπει η αντίδραση να είναι ταχεία θα ε, σταματήσουν οι δασμοί για 75 κατηγορίες προϊόντων. Βρίσκω ότι είναι σωστή η βοήθεια αυτή προς το Πακιστάν. Βέβαια, όπως είπα και τονίζω και πάλι, ότι χρειάζεται ταχεία αντίδραση. Δεν πρέπει να διαρκέσει πολύ, γιατί το Πακιστάν χρειάζεται τώρα την ε, οικονομική αυτή ενίσχυση, όχι σε ένα χρόνο. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν σημαντικές αντιστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ε, βιομήχανοι κλωστοεφαντουργικών προϊόντων ε, θα εκστρατεύσουν κατά της διευκόλυνσης αυτής εισαγωγών τέτοιων προϊόντων από το Πακιστάν. Αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας σταματήσει αυτό, διότι χρειάζεται, όπως είπα, ταχύτατη αντίδραση. Ο Ευρωπαίος καταναλωτής πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη. Περί αυτού πρόκειται. Να δείξουμε ότι και για μας έχει αξία η επίδειξη αυτή αλληλεγγύης διότι δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία να ταχθεί κανείς υπέρ της, του ελεύθερου εμπορίου από ότι σε αυτή την πρόταση. Τώρα είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι. Ας προσέξουν να μιλήσουν για ένα λεπτό ο καθένας, όχι παραπάνω, για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Η κυρία Κόμου πρώτη θα πάρει το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με τη σύντομη αυτή παρέμβασή μου θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη άρση φόρων στο Πακιστάν για διάστημα ε, τριών ετών για 74 προϊόντα που αφορούν τον τομέα τη ένδυση και τη φιλοστοφαντουργία. Ο προβληματισμό μου αφορά τι αρνητικέ επιπτώσει τη ευρωπαϊκή βιομηχανία και ιδιαίτερα τη Ιταλική και ε, στην πόλη απασχόλη στην Ευρώπη σε ένα τομέα που πλήττεται από την οικονομική κρίση. Ιδιαίτερα σκέφτομαι τι μικρομεσαίε επιχειρήσει του τομέα που προσπαθούμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και που δίχω άλλο θα υποστούν ένα σοβαρό πλήγμα. Δεν είναι ασήμαντο το γεγονό ότι το Πακιστάν επέβαλε με ένα φόρο 15% στις εξαγωγές ε, κλωστών ε, ε, βαβακερών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τις πρώτες ύλες προσπαθώντας, προσπαθεί να διατηρήσει ένα χαμηλό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι η χώρα αυτή επλήγει από καταστροφές. Η ευρωπαϊκή χώρα που μπορώ να φανταστώ είναι να συμβάλλει στη δημιουργία υποδομών και δρόμων χρησιμοποιώντας το τοπικό εργατικό δυναμικό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι εύκολο να συζητήσει κανείς αντικειμενικά όταν γνωρίζει ότι 100.000 παιδιά έχουν μείνει άστεγα, ότι εκατομμύρια αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και νομίζω ότι είναι σωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει γρήγορα. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι τα μέτρα που προτείνεται βοηθούν άραγε σωστά ή βοηθούν τους λάθος ανθρώπους. Εδώ θα πρέπει να το εξηγήσετε λίγο καλύτερα. Διότι είναι δικαιολογημένο να πει κανεί ότι στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας βοηθεί μεν το σύνολο του Πακιστάν, αλλά δεν γνωρίζω αν η βοήθεια πραγματικά θα καταλήξει στα χέρια των ανθρώπων που τη χρειάζονται περισσότερο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι εάν αυτή η βοήθεια σημαίνει ότι θα μπορέσει να αυτοβοηθηθεί το Πακιστάν, τι συνέπειε, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην Ευρώπη. Όντως οφείλουμε να βοηθήσουμε. Ελπίζω όμως ότι με την βοήθεια αυτή θα βοηθήσουμε πραγματικά τα πρόσωπα εκείνα που την έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λάμπερτ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να απαντήσω σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που υπευλήθησαν. Αυτό που θα τώρα να κάνει το Πακιστάν είναι να βοηθήσει εαυτόν για να γλιτώσει αυτά τα προβλήματα της κοινωνικής καθολικής πλημμύρες και βέβαια ευτυχώ τα εργοστάσια δεν είναι στις περιοχές που επλήγησαν. Ε, βέβαια η άμεση βοήθεια σε σχέση με τις ανάγκες δεν είναι τίποτα, είναι πενταροδεκάρες η κατανομή του εισοδήματος από τις επιπλέον εξαγωγές είναι κάτι το σημαντικό υποδομές, ενέργεια, παιδεία, ε, δρόμοι και βεβαίως ε, την ευθύνη τώρα την έχει η δημοκρατική, ε, δημοκρατία κλεγμένη κυβέρνηση σε σχέση με φορολογικά έσοδα κλπ. Εάν υπήρχε περισσότερη πολυμορφία στην βιομηχανία, αν δεν ήταν τόση συγκέντρωση στα κλωστοματουργικά θα είχε άλλωση, η όλη προβληματική. Όμως να η ευκαιρία που έχει αυτή η χώρα και ευκαιρία που έχουμε εμεί να τους βοηθήσουμε να γλιτώσουμε αυτή την καταστροφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κατάσταση στο Πακιστάν απαιτεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν θα πρέπει όμω να είναι πρόφαση για να πληγεί η παντουργία των χωρών μελών όπω τη Πορτογαλία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να είναι κανεί αλληλέγγυος με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, πιο άμεσο που θα βοηθήσει τις πληγήσεις περιοχές. Υπάρχουν πιο σωστοί τρόποι βοήθειας προτάσεις αυτές ε, δεν είναι καλές μακροπρόθεσμα. Στην ουσία μόνο, είναι μόνο υπέρ ε, λίγων και για λίγο χρονικό διάστημα την, ε, η κλωστοφαντουργία πλήττεται από την άλλη. Σε ένα πλαίσιο κρίσης και ανεργίας οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν πρόφαση για απολύσει. Βεβαίως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ε, συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού. Ο κοινοτικό προπολογισμό προβλέπει ένα κονδύλιο για τη δημιουργία ενό κοινοτικού προγράμματο για την υποδοματοποιία και την γλωσσοφαντουργία. Ήμασταν εμεί αυτοί που το ψηφίσαμε. Πού κατέληξε αυτό το κονδύλιο, τι μπορεί να μα πει ο ε, Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι παράδοξο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να υπερασπιστεί τι δικέ μα θέσει εργασία, τι διακυβεύει πίσω από την ρητορική των, ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας η μείωση των φόρων για τα επόμενα τρία χρόνια και προϊόντα ένδυσης που προέρχονται από το ε, Πακιστάν υπάρχει κίνδυνος να καταβαραθρώσει το τομέα της ε, μεταποίησης με απώλεια θέσεων εργασίας. 40.000 από τις θέσεις εργασίας που θα είναι στην Ιταλία. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε εμπορικά μέτρα όταν στη χώρα μας και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχουν προβλήματα από τις ασιατικές χώρες και κυρίως από την Κίνα. Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει φιλανθρωπία εις βάρος της Ιταλίας που αντιπροσωπεύει το 30% του ευρωπαϊκού κουρστοφεντουργικού τομέα. Ζητώ παράλληλα με το Πακιστάν να βοηθήσουμε και τις δικές μας μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση επιβάλλοντας φόρους στα ασιατικά προϊόντα. Είμαι από το Πράτο και εμείς ε, πραγματικά οι κάτοικοι του Πράτο έχουμε ε, φτάσει το ε, ε, σε ένα σημείο κορεσμού. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την μεταποιητική βιομηχανία, θυμίζω ότι το Πακιστάν αποτελεί παγκοσμίω τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό βάμβακος με ποσοστό 9% της παγκόσμιας παραγωγής, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έπεται με μόλις 5,5%. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό Βεβαίω δεν θέλουμε προστατευτισμό που θίγει τον υγιή ανταγωνισμό. Θέλουμε ελεύθερο και ανοιχτό διεθνέ εμπόριο. Απ' την άλλη όμω αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι, ένα πολύ παραστατικό ο κύριο Μέλο, ε, που προέρχεται και από μια χώρα με ευαίσθητη οικονομία την πορτογαλία. αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στην ιταλία προσθέτω και εγώ την ελλάδα που ξέρετε όλοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. βεβαίω να ενισχύουμε το πακιστάν να ελέγξουμε όμω και αυτό ε, θέλω να ρωτήσω την επιτροπή κατά πόσο έχουμε του μηχανισμού που διασφαλίζουν ότι οι ενισχύσει που ε, ε, δίνουμε στο πακιστάν κατευθύνονται σωστά και δεν χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση άλλων σκοπών και κάποιων βιομηχανιών σε βάρος ευρωπαϊκών ε, εταιριών και ευρωπαίων εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, ο κύριος το λόγο τώρα θα πάρει. Δεν είμαι εμπειρογνώμονα τα σχετικά θέματα, όμως είναι σοβαρό το θέμα, είναι σοβαρή χώρα το Πακιστάν, που δεν έχει ποτέ σταθερό καθεστώς, που είναι σε περιοχή τόσο ασταθή, όπως ο κύριος Καρύμ. Εμείς μια που έχουμε την ευημερία και την ειρήνη θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στο να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό στον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως δεν μπορώ παρά να υποστήριξω τη σημερινή πρόταση. Όμως παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας απαντήσει σε αυτά τα θέματα ε, διότι θα πρέπει να παρασχεθούν κάποιες εγγύσεις ότι η ενίσχυση θα φτάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται και δεν θα πάει στους γεωκτήμονες και στους ε, κερδοσκόπους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν προκάλεσαν ε, βαρύτατες ε, συνέπειες ε, για τους ανθρώπους εκεί. Μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας του Πακιστάν έχουν λοιπόν ζωτικό χαρακτήρα. Θεωρώ όμως αμφισβητούμενο εάν απλή μείωση των δασμών θα επιτύχει τον στόχο αυτό. Υπάρχει κίνδυνος έμεσα να επωφεληθούν τρίτες χώρες και έτσι να μην επιτευθούν οι επιθυμούμενοι στόχοι. Η συγκεκριμένη ερώτηση που υποβάλλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εάν η μείωση των δασμών της εθανόλης πραγματικά θα ωφελήσουν τους ανθρώπους στο Πακιστάν και αν μπορεί να υπολογιστεί εάν διατηρούνται πραγματικά συνθήκες βιωσιμότητας της παραγωγής εθανόλης στο Πακιστάν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Σιλβέστρης έχει, θα πάρει το λόγο, αλλά προηγουμένως νομίζω να, θέλει να παρέμβει ο κύριος Ντάτμουρ. Ναι, έχετε το λόγο. Αναρωτιέμαι αν συνειδητοποιείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε τις ενισχύσεις, συζητάμε εμπορικές προτιμήσεις και αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο Πακιστάν να επιλύσει τα προβλήματά του μόνο του. Ελπίζω ε, να το συνειδητοποιείτε αυτό. Ε, Νομίζω ότι αυτό είναι το θεμελιώδες ε, στοιχείο της ε, απόψινής συζήτησης τα μέτρα λοιπόν πρέπει να είναι καλά μελετημένα ώστε να δώσουν με βιώσιμο τρόπο μια ενίσχυση. Και για το λόγο αυτό είναι σημαντική και μια λύση κόστους και ωφέλους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεχίζουμε ο κύριος Σιλβέστρης τώρα θα πάρει το λόγο. Διαδικασία κάτσου διάρρη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Presidente, non vi è dubbio. Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ανάγκη παρέμβαση μετά από τι πλημμύρε που έπληξαν το Πακιστάν. Σήμερα όμω θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι το είδο τη ενίσχυση που χρειάζεται περισσότερο αυτή η χώρα και ποια είναι η ενίσχυση που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δράσουμε ταχαίω, αλλά να είμαστε και αποτελεσματικοί. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, εγώ τρέφω σοβαρέ αμφιβολίε. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια πρόταση που έχει πάρα πολλά και υπάρχει ο κίνδυνο παρεμβαίνοντα στον τομέα τη βιωσιοδεψία και τη κλωστοφαντουργία να μην είναι επαρκώ αποτελεσματική. Πιστεύω ότι θα δημιουργήσει πολύ περισσότερε εντάσει και θα γονατίσει τον τομέα αυτό στην Ευρώπη, ένα τομέα που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ύστερα το να ευνοήσουμε τι εξαγωγέ από πλευρά επιχειρήσεων που παράγουν σημαίνει ότι βοηθάμε τι χώρε, τα μέρη εκείνα στο Πακιστάν που δεν έχουν πληγεί από τις ε, πλημμύρες. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες να ξεκινήσουν και πάλι την παραγωγή. Πιστεύω ότι η οδό τη εξάλληψη των φόρων είναι ο πλέον ακατάλληλος δρόμο, ε, ο οποίος δεν μας βρίσκει που δεν είναι σύμφωνο. Ευχαριστώ. Τελείωσαν οι παρεμβάσει των βουλευτών και η συζήτηση θα κλείσει με τον κύριο Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, θα πάρετε το λόγο. Thank you. Um, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, να διατυπώσω σαφώς περί ομιλούμε, περί τι ποσόν ομιλούμε. Μιλούμε για ένα όγκο συναλλαγών της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα θα είναι λοιπόν αύξηση των εξαγωγών του Πακιστάν προς την Ένωση της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι ίδιες οι εισαγωγές, το συνολικό ισοζύγιο δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μοναχά 50 εκατομμύρια. Διότι λόγω της πιο ευνοϊκής θέσης του Πακιστάν να εξάγει προς την ευρωπαϊκή αγορά, θα υπάρχει και μία διαφοροποίηση των ε, εμπορικών ροών Άρα ορισμένοι θα υποφεληθούν από τις ροές αυτές στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή μιλούμε για περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το λέω αυτό γιατί άκουσα πάλι στην απόψινή συζήτηση ότι θα χαθούν 120.000 θέσεις εργασίας. Στα κινητά σας τηλέφωνα όλοι έχετε έναν μικρό υπολογιστή. Για να χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 120.000 θέσεις εργασίας μόνο από αύξηση 50 εκατομμυρίων ε, ευρώ, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ προβληματική η ευρωπαϊκή η βιομηχανία. Δεύτερο, λάβαμε δεόντως υπόψη τις ευαισθησίες της ευρωπαϊκής υφαντουργίας. Και λάβαμε επίσης υπόψη την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η ε, βιομηχανία αυτή. Δεν είναι λοιπόν ε, ούτε τα λινά τμήμα της συμφωνίας, ούτε ε, ορισμένα είδη ενδύσεως. Και αυτά είναι σημαντικά για την Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, περιλαμβάνονται πολλά ημιέτοιμα προϊόντα. Όταν λέμε ημιέτοιμα προϊόντα, σημαίνει ότι θα ολοκληρωθούν, θα τελειοποιηθούν στην Ευρώπη. Άρα, θα είναι Φθηνότερε οι εισαγωγέ υπέρ των ε, βιομηχανιών εκείνων οι οποίε θα τελειοποιήσουν τα προϊόντα. Άρα αυτό δεν μα βλάπτει άμεσα, αντίθετα μάλιστα μα ωφελεί. Έχουμε λοιπόν μελετήσει ε, με μεγάλη ακρίβεια μια πρόταση η οποία θα ωφελήσει το Πακιστάν χωρίς να βλάψει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σε μια περίοδο βέβαια που εξερχόμαστε από μια κρίση και που σίγουρα η οικονομία δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Έγινε μια παρατήρηση επίσης σχετικά με τις εξαγωγές βαμβακιού. Σε ολόκληρη την παγκόσμια αγορά υπάρχει μια σπάνης βαμβακιού και βέβαια το Πακιστάν είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βαμβακιού. Αυτό που έχω υπόψη είναι αυτή τη στιγμή κυρωθεί η συμφωνία αυτή και μπορούμε κάπως να προχωρήσουμε. Νομίζω πρέπει να ζητήσουμε από το Πακιστάν να εξασφαλίσει ώστε και η δική μας η βιομηχανία να έχει αρκετό βαμβάκι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Αφού όπως είπα υπάρχει ε, έλλειψη βαμβακιού παγκόσμια για ορισμένα είδη βαμβακιού τουλάχιστον ορισμένες ποικιλίε βαμβακιού ε, διότι ε, και οι αφρικανικές χώρες παράγουν πολύ βαμβάκι δεν παράγουν πάντοτε τα είδη εκείνα που χρειαζόμαστε και ούτε μπορούν να αλλάξουν την παραγωγή τους από την μια μέρα στην άλλη. Έτσι λοιπόν έχουμε λάβει και υπόψη, υπόψη και αυτό το ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε λέγοντας ότι νομίζω ότι όταν εξετάζει κανείς την κατάσταση του Πακιστάν αυτό που χρειάζεται η χώρα αυτή είναι και περισσότερη βοήθεια αλλά και περισσότερο εμπόριο. Χρειάζεται και τα δύο λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ήδη 320 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια. Είναι περίπου το 60% αυτών που ζήτησε τα Ηνωμένα Έθνη. Το trade δεν σημαίνει aid. Το εμπόριο δεν είναι απλή ε, βοήθεια. Το εμπόριο σημαίνει να δοθούν ευκαιρίες στην ε, ισπανική βιομηχανία για να αυξήσει τις εξαγωγές της και να δώσει δουλειά στους ανθρώπους που την χρειάζονται επιτόπου. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό εργαλείο για την ανάκαμψη της οικονομίας τους, να τους προσφέρουμε και άλλες εμπορικές δυνατότητες δεν μιλούμε ειδικά για βοήθεια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα ωφεληθούν από αυτό είναι βέβαια πολύ πιο εύκολο να γίνει με την άμεση παροχή βοήθειας. Δεν μπορεί όμως κανείς να στηρίξει τα πόδια της μια οικονομία μόνο με παροχή άμεσης βοήθειας. Γι' αυτό χρειάζεται και η βοήθεια αλλά και ε, το εμπόριο. Ας μην λησμονούμε, όπως είπα ήδη ενώπιον σας, ότι μιλούμε για μια περιοχή του κόσμου η οποία επλήγει βαρύτατα. Ένας Ιταλός ευρωβουλευτής στην παρέμβασή του ε, συνέ... Ε, ε, λέω εγώ ότι μπορεί να συγκρίνει κανείς την περιοχή που έχει πληγεί από τις πλημμύρες στο Πακιστάν είναι περίπου τόση σε έκταση όσο η Ιταλία. Το Πακιστάν είναι πολύ σημαντικό στρατηγικά και για μας, για την ασφαλειά μας. Θα ήταν λοιπόν πολύ επικίνδυνο για την Ευρώπη εάν η περιοχή αυτή γίνει ασταθής. Πρέπει λοιπόν να πράξουμε πάντο δυνατόν ώστε ε, να συμβάλλουμε στη διατήρηση της σταθερότητας της περιοχής αυτής. Πρόκειται λοιπόν για ένα φάσμα μέτρων. Ε, συνεχίζουμε τις πολιτικές συζητήσεις με το Πακιστάν, ε, πρόσφατα σε διάσκεψη κορυφής με τους ηθήνοντες της χώρας αυτής. Επίσης, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μετέβησαν εκεί. και η Επίτροπος Γεωργίευα για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε και την δέσμη μέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας πολύ σημαντική. Έχουμε και μια οικονομική προσέγγιση που σημαίνει επομένως περισσότερο εμπόριο με την χώρα αυτή. Ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό βοηθούμε σημαντικά την χώρα αυτή. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι βοηθώντας το Πακιστάν βοηθούμε και τους αυτούς μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έληξε η συζήτηση για αυτό το θέμα και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της κυρίας Μουσκαρντίνη με θέμα ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα